στην ψηφοφορία. Έχουμε τρεις προτάσεις για την Ικαράγουα. Έχει ζητήσει το λόγο η Ντεκεζέρ. Η ομάδα μας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ψηφοφορία για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως ούτε αποχή καν απλώς δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία. Κύριε Κορχολά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτηση ήταν πάρα πολλοί οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεπεράσουν το χρόνο αγορευσής τους. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αν είναι απαραίτητο μπορείτε να τους κόβετε και το μικρόφωνο καμιά φορά. Είναι σημαντικό για να μην χάνουμε τόσο χρόνο αγόρευσης χωρίς λόγο. Ορισμένοι λέει ο πρόεδρος. Είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν δύο φορές, αλλά ή, όχι για το ίδιο σημείο. Εγώ δεν εμπόδισα κανένα να περάσει το όριο, την επόμενη φορά όμως θα το πράξω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Και εγώ θέλω να τονίσω το γεγονός ότι και η δική μας ομάδα, όπως και οι σοσιαλιστές, δεν θα συμμετάσχουμε στη ψηφοφορία και θέλουμε να καταγραφεί η στάση μας και στη συζήτηση και στην ψηφοφορία. Κυρία Φιγκερέντου, χωρίς, χωρίς μικρόφωνο. Και εμείς έχουμε ακριβώς την ίδια κατεύθυνση για τους λόγους που εξηγήθηκαν προηγουμένως από τη, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών μας. Δεν θα συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία. Προφανώς λάβαμε μέρος στην συζήτηση, αλλά δεν θα λάβουμε χώρος στην, ε, στην ψηφοφορία που δεν είναι πραγματικά κατεπήγον θέμα όπως τονίσαμε στην, στην ε, παρέμβασή μας. Dobře, děkuji. Ja myslím, że můžeme přistoupit k hlasování. o Θα ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα του ΕΛΚ, των Φιλελευθέρων και των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών για την Ικαράγουα. Ποιος είναι υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στο δεύτερο σημείο που είναι η, ψηφοφορία τεσσάρων ψηφισμάτων για το Βιετνάμ και το Λάος. Παρακαλώ. Υπήρξε ένα μικρό τεχνικό λάθος. Εκεί που αναφέρεται πειθαρχική και ποινική, οι δύο όροι πειθαρχικός και ποινικός θα διαγραφούν. Για το Λάος και το Βιετνάμ, κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων. Παρακαλώ. Παράγραφος 6. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Προκύ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολόκληρο το ψήφισμα τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα. Τέλος, έχουμε την ψηφοφορία πέντε ψηφισμάτων για την Κίνα, την, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Ο κύριος Πόσελ ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα λάθος στο σημείο 3 στο γερμανικό κείμενο και θα ήθελα να το κοιτάξουμε εκεί και να το διορθώσουμε και στα γερμανικά και στις άλλες ε, μεταφράσεις ότι αναφέρεται ότι η εκτέλεση των δύο Θιβετιανών καθώς και εννέα άλλων Ουιγούρων. Αυτό δεν ισχύει γιατί οι Ουιγούροι δεν είναι Θιβετιανοί ούτε το αντίστροφο. Λοιπόν, να διορθωθεί παρακαλώ σε όλες τις γλωσσικές εκδοχέ. Ευχαριστώ κύριε Πόσελ, τι λέει ο Πρόεδρος, θα το διορθώσουμε. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία του ψηφίσματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα το κοινό ψήφισμα τριών πολιτικών ομάδων. ΕΛΚ, Φιλελευθέρων και Πρασίνων. Ψηφίζουμε παρακαλώ ονομαστικά. Ή μάλλον την παράγραφο 9 λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Λάθος, λάθος. Παράγραφος 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ετοιμάστε παρακαλώ τις κάρτες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Τέλος ψηφοφορίας παρακαλώ. Το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται η παράγραφος 9. Τώρα ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Οπότε διακόπτουμε τη σύνοδο μέχρι την επόμενη ολομέλεια. Μια και δεν υπάρχουν, ε, αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ε, για τα πρακτικά, θα, μεταβλη, ε, διαβιβαστούν τα έγγραφα σε όλα τα θεσμικά όργανα που αναφέρονται, αναφέρονται στο, στην ημερήσια διάταξη. Διακοπή τη